επεξηγήσεις ψήφου, αλλά θα ήθελα πρώτα να ζητήσω από τους συναδέλφους να φύγουν από την αίθουσα χωρίς θόρυβο. Λοιπόν, συνάδελφοι, ακολουθούν επεξηγήσεις ψήφου τώρα. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο Ματ Κάρθι, τον οποίο δεν βλέπω. Α, όχι, σας βλέπω. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Συγγνώμη, μην αρχίζετε ακόμα. Παρακαλώ, συνάδελφοι, να ακούσουμε λίγο τις επεξηγήσεις ψήφου. Ησυχία.

ευκαιρία να ε, προστατεύσουμε τις ε, προδιαγραφές και το καθεστώς χωρών όπως η Ιρλανδία ως προς τα μεταλλαγμένα. Θα μπορούσε να είναι προς το καλύτερο συμφέρον των πολιτών. Αντί να γίνουν όλα αυτά, στράφηκε προς τα συμφέροντα των βιοτεχνολογικών εταιριών. Εμείς και άλλες πολιτικές ομάδες δεν ε, πέσαμε στον πειρασμό να περάσουμε ε, γρήγορα μια τέτοια νομοθεσία. Εμεί από το Συνφέιν και κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να ανεχθούν μια τέτοια νομοθεσία που αφήνει παραθυράκια επικίνδυνα. Ε, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μπόιλαν που ήταν σκιώδη συγγήτριά μα και εξήγησε τη θέση τη συντριπτική πλειονότητα Ιρλανδών και άλλων Ευρωπαίων πολιτών. Θα εξακολουθήσουμε να πιέζουμε για απόλυτη σαφήνεια τα κράτη-μέλη να μπορούν να ε, απαγορεύουν αυτές οι καλλιέργειες προς όφελος των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και τοπικών κλάδων της οικονομίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ποσπίσιλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ χαιρετίζω τον συμβιβασμό διότι είμαι πεπισμένος ότι αντιπροσωπεύει λύση λύση που δεν ικανοποιεί ούτε τους υπέρ ούτε τους κατά απόλυτα αλλά επιτρέπει στα κράτη-μέλη να απαγορεύουν την καλλιέργεια μεταλλαγμένων στην επικράτειά τους και αυτό νομίζω ότι είναι σωστό. Μια συγκεντρωτική θέση που θα επέβαλε στα κράτη-μέλη την καλλιέργεια ή μη των μεταλλαγμένων σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν θα ήταν σωστή γιατί θα παραβίαζε την κυριαρχία των χωρών μελών. Η θέση της τσεχικής δημοκρατίας που προσωπώ εδώ είναι και ήταν ότι το κατά πόσον τα κράτη-μέλη θα επιτρέψουν ή όχι την καλλιέργεια μεταλλαγμένων πρέπει να είναι δικό τους θέμα και πιστεύω ότι ο συμβιβασμός αυτός είναι πολύ σωστός. Ευχαριστούμε. Μπόγκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ. Υποστηρίζω την πρόταση και αυτό διότι διορθώνει μία κατάσταση που είχε δημιουργηθεί από χρόνια όταν ήμουν υπουργό Γεωργίας και θυμάμαι τι έλεγαν τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο. Μερικά από αυτά ήταν ομά και προσπαθούσαν να πιέσουν ομά για, την, ε, για να επιτραπεί η καλλιέργεια των μεταλλαγμένων. Ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν σε αυτόν τον συμβιβασμό και τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας μεταξύ άλλων. Γνωρίζουμε τι λέει ο συμβιβασμός. Τα κράτη-μέλη μπορούν να πάρουν την απόφαση χωρίς να ε, μηνυθούν από πολυεθνικές εταιρείες. Μπορούν να δεχτούν ή μη την καλλιέργεια των μεταλλαγμένων. Επίσης σημαντικό είναι ότι η συμφωνία αυτή εγκρίθηκε και από το Κοινοβούλιο πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Σημαντικό. Κύριο Ζάχαντρα για ένα λεπτό. Ζάχαντριλ. Ζάχαντιλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ χαιρετίζω το αποτέλεσμα. Ψήφισα και εγώ υπέρ για δύο λόγους. Διότι πρώτον είναι καλό να μπορούν τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν τα ίδια όπου δεν χρειάζεται να νομοθετήσει η Ένωση. Και εδώ ακριβώς, για αυτή την περίπτωση ακριβώς πρόκειται. Δεύτερον, σε μερικές χώρες μέλη υπάρχει μία ιστερία, αντιεπιστημονική ιστερία κατά των μεταλλαγμένων δεν νομίζω ότι παραβιάζω την άποψη καθενός αν πω ότι έχει το δικαίωμα όποιος δεν θέλει μεταλλαγμένα να μην τα καλλιεργήσει αλλά δεν πρέπει να υποχρώνονται οι υπόλοιπε χώρες να ακολουθήσουν. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αυτή η απόφαση θα ξεμπλοκάρει το βέτο που ισχύει αυτή τη στιγμή πανενωσιακός. Εάν πράγματι θέλουμε εμείς να καλύψουμε τις τροφιμικές ανάγκες του πληθυσμού και να καταπολεμήσουμε τις ασθένειες λόγω του κλίματος, θα πρέπει να ελέγξουμε τις επιστήμες στον τομέα της παραγωγής προϊόντων. Η κατάσταση αυτή, η ακινησία στα γενετικά τροποποιημένα κράτησε πάρα πολλά χρόνια και γι' αυτό υποστηρίζω την συγκεκριμένη απόφαση η οποία λύνει τα χέρια των κρατών μελών. Η περιφέρεια που εκπροσωπώ έχει κάποιες από τις καλύτερες καλλιέργειες στον κόσμο. Ε, στο Κέμπριτζ όπου στις περιοχές όπου παράγονται πατάτες οι οποίες δεν υποφέρουν από συγκεκριμένες μορφές ασθένειας μπορούν τα προϊόντα αυτά να χρησιμεύσουν στη διατροφή του προϊόντος, του πληθυσμού. Θα έπρεπε να υπάρχει λοιπόν μια λύση η οποία να βασίζεται σε αποκλειστικά επιστημονικά στοιχεία. Λόγω όμως της κατάστασης αυτής της τασιμότητας τόσα χρόνια πρέπει να δώσουμε την δυνατότητα και στην επιστήμη και στις χώρες να προχωρήσουν. Τζάλκ. Ο τριμερής διάλογος από τις 3 μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου είναι μια κατελάχιστον συμφωνία που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να καλλιεργούν γενετικά τροποποιημένα εφόσον το επιθυμούν. Ε, δεν πρέπει να έχουμε όμως ψευδεστήσεις. Δεν έχουμε να κάνουμε με μια πρώτη φάση εθνικού τύπου ανταπάντησης στις προτάσεις για τα γενετικά τροποποιημένα, αλλά πρόκειται για μια θα έλεγα φιλανθρωπία την οποία κάνουμε προς τα κράτη-μέλη τίποτα δεν λέγεται για τη δυνατότητα που πρέπει να έχουν τα κράτη-μέλη να ε, επιβάλλουν την σήμανση των προϊόντων ε, που περιέχουν ε, γενετικά τροποποιημένα. Απαγορεύουν την καλλιέργεια στα εδάφη τους και εισάγουν προϊόντα τα οποία είναι γενετικά τροποποιημένα. Είμαστε στην ουσία στα χέρια ισχυρών επιχειρήσεων οι οποίες ελέγχουν τη γενετική επιστήμη εις βάρος της υγείας, ενώ αλλού οι συζητήσεις και οι πολίτες μετέχουν και στη Ρωσία μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Λούνατσεκ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Εκατομμύρια ήταν και παραμένουν οι πολίτες, άνδρες και γυναίκες καλλιεργητές βιολογικών, καταναλωτές στην κοινή μας Ευρώπη που μετά από χρόνια εμπλοκής ε, στο Συμβούλιο και μεγάλες αντιστάσεις στις πολυεθνικές κατέστησαν δυνατή τη σημερινή επιτυχία. Δεν λέω, συμβιβασμό είναι, αλλά είναι μια σημαντική πρόοδο και ένα βήμα πρόοδου. Με τη δική μου υπερψήφιση σήμερα, εγώ θέλω να δείξω σε όλου όσοι ενδιαφέρονται, στι οργανώσει περιβαλλοντικέ, ότι υπάρχουν 62 περιφέρειες στην Ευρώπη και θέλω να τις ε, σεβαστώ και να ποτίσω ένα φοροτιμής. Και αυτό ξεκίνησε από την Άνω Αυστρία πριν από 11 χρόνια σε αυτό το ομοσπονδιακό κράτος της Αυστρίας. Τι να κάνουμε, είναι μισοάδιο το ποτήρι ε, ε, και μισογεμάτο με ένα, αλλά λείπουν ακόμα μερικά στοιχεία είναι απαράδεκτο να δίνετε δικαίωμα λόγου στις πολυεθνικές εταιρείες και χρειάζεται πιο δημοκρατική διαδικασία έγκρισης. Αυτό μας το έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος Ιούνκερ και έχει αναθέσει στον Επίτροπο Ανδρουκάητης μέχρι αρχές Μαΐου να φέρει νέα πρόταση. Αυτό οπωσδήποτε πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ η κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ ψήφισα αποχή για αυτή την πρόταση οδηγίας. Διότι παρά τη βελτίωση του κειμένου, δεν είναι αρκετή η προστασία της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών, ούτε ε, η επικορικότητα. Το είπα και προηγουμένως. Ε, έχουμε ευθύνη για τα τρόφιμα και έχουμε ευθύνη και για τη βιοπικιλότητα η γενετική τροποποίηση μπορεί να έχει επιπτώσεις και στην ανθρώπινη υγεία αλλά και στο περιβάλλον. Οι εταιρείε ε, αυτές ε, της γενετικής τροποποίησης και γενετικής τεχνολογίας θέλουν η Ευρώπη να είναι ξέφραγο απέλη. Εμείς θελήσαμε να τους δείξουμε ότι τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που αποφασίζουν. Δεν καταφέραμε όμως να προστατευτούμε από τις εταιρείε αυτές ούτε από τη ρήπανση του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να παραμείνει πράσινη ήπειρος. Ελπίζω η Επιτροπή Γιούνκερ να φέρει όντως νέα πρόταση οδηγίας που θα είναι πιο πράσινη, πιο οικολογική κατά το μεταλλαγμένο. Ευχαριστώ κύριε Κινίτσι. Madame, you have Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων προκαλεί τεράστιες συζητήσεις όχι μόνο στο εσωτερικό των κρατών μελών αλλά ε, και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινή γνώμη ε, έχει διαρρεθεί διότι δεν είναι ξεκάθαρη οι συνέπειες στην υγεία των πολιτών. Μετά από τρία χρόνια διαπραγματεύσεων το κείμενο καταλήγει σε μια ισορροπημένη συμφωνία που σέβεται την αρχική συμφωνία του 2001 δίδοντας μεγαλύτερη νομική ασφάλεια στις δυνατότητες των κρατών μελών να περιορίσουν εν μέρη ή συνολικά στο έδαφος τους την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων. Παραμένει λοιπόν η ελευθερία επιλογής εκτιμώντας τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τους κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων όπως επίσης και τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις στην γεωργία. Η συμβιβαστική αυτή λύση είναι μια καλή λύση, διασφαλίζει την υγεία του καταναλωτή κυρίως και γι' αυτό θα την υπερψήφισα. Ευχαριστώ η κυρία Γκαρντίνη. Ε, υπερψηφίσαμε την πρόταση αυτή η οποία ήταν σε αναμονή θα έλεγα εδώ και τρία χρόνια και πράγματι επιτρέπει στα κράτη-μέλη να επιτρέψουν ή να απαγορεύσουν τα γενετικά τροποποιημένα στα εδάφη τους. Η βασική αρχή εδώ είναι η αρχή της επικουρικότητας, ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που αφορά την περιβαλλοντική ασφάλεια και την τροφιμική ασφάλεια. Η μεγάλη στήριξη την οποία έλαβε η πρόταση αυτή από όλες τις πολιτικές ομάδες σχεδόν δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ευαίσθητο απέναντι στους πολίτες που θέλουν να διοτηρήσουν τα θεμέλια μιας γεωργίας με υγεία και ασφάλεια. Ε, υπάρχει ένα θέμα εδώ της οικονομικής ευθύνης, εξαιρέθηκε από την πρόταση και θα πρέπει να μας απασχολήσει γιατί νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι οικονομικές βλάβες μπορεί να προκληθούν από τις γενετικά τροποποιημένες στις γειτονικέ καλλιέργειες και ποιος θα καλύψει τις ζημίες αυτές οικονομικά. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Τζούφριντα. Ευχαριστώ. Όλοι γνωρίζουμε ότι το θέμα των γενετικά τροποποιημένων είναι ένα θέμα που ενθουσιάζει και δημιουργεί τεράστιες συζητήσεις και ξέρουμε ότι η κοινή γνώμη είναι κατά 58% κατά. Βέβαια φαίνεται εδώ ότι υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία είναι η επιστημονική άποψη, την οποία εκφράζουν οι λεγόμενοι σε εισαγωγικά κακοί, ε, και στην συναισθηματική αντίληψη η οποία είναι η λεγόμενη καλή ή η άποψη των καλών που φοβούνται την πρόοδο. Νομίζω ότι οι διαφωνίες υπάρχουν κυρίως στον επιστημονικό κόσμο. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις από τις επιστήμες. Δεν έχει αναπτυχθεί δυστυχώς μία μη ιδεολογική συζήτηση στον τομέα της επιστήμης γύρω από αυτά. Ο κάθε ένας βουλευτής λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσει να ευαισθητοποιήσει τις χώρες του για να υπάρξει έρευνα, να υπάρξει αναζήτηση. Είναι μια καλή πρόταση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν μου αρέσει πάρα πολύ και εμένα ο συμβιβασμό, παρόλα αυτά τον υπερψήφισα. Διότι αντανακλά την πολιτική πραγματικότητα αλλά και μας ανοίγει μια νέα διαδικασία. Δεν μπορούσε να συνεχιστεί η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και το Συμβούλιο είχαν αλληλοδηγηθεί σε εμπλοκή. Τουλάχιστον προσπαθούμε λίγο να προχωρήσουμε. Έχω μια επιθυμία μόνο. Παρ' όλα αυτά να προχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τομέα της γενετικής τεχνολογίας, κυρίως σε ό,τι αφορά την εκτίμηση κινδύνου, να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ πιστεύω ότι το να είσαι απλώς κατά δεν βοηθάει. Καλύτερα να έχουμε επιστημονικές μελέτες και να συμμετέχουμε στην εκτίμηση και αξιολόγηση του κινδύνου και με τη νέα διαδικασία αυτό καθίσταται δυνατό. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Γκόλιν για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το κείμενο που έχουμε ενώπιόν μας είναι δούριος ύπος γιατί την πρόφαση ότι δίνει ελευθερίες ε, στη κράτη-μέλη ε, θέτει τους ε, αγρότες όμοιρους στα χέρια των πολυεθνικών. Γνωρίζουμε ότι βλάπτει αυτή η κατάσταση τη χλωρίδα και την πανίδα. Είναι απαράδεκτα. Μας αλυσοδένει ακόμα περισσότερο στην παγκοσμιοποίηση και στην ειδίκευση των καλλιεργειών. Χάνουμε τις ιδιαιτερότητες και της διατροφής και του τοπίου μας. Για να υπηρετήσουμε ποιους, όχι τους λαούς, αλλά τους μετόχους κάποιων εισηγμένων εταιριών. Ε, λένε ότι δεν μπορούμε να ταΐσουμε την ανθρωπότητα χωρίς ε, ε, μεταλλαγμένα. Δεν ισχύει αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε τις σωστές πολιτικές επιλογές. Το κείμενο αυτό είναι αντίθετο με οποιαδήποτε ε, επισητιστική κυριαρχία που για τους λαούς είναι ό,τι και ελευθερία για το άτομο. Θα πρέπει να αποφασίζουμε τι θέλουμε εμείς να τρώμε και να τρώνε τα παιδιά μας χωρίς κινδύνους για την υγεία. Ε, γι' αυτό εγώ καταψήφισα το κείμενο αυτό. Ο κύριος Άνεμανς, για ένα λεπτό παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η βελτίωση των ειδών δεν γίνεται μόνο με τη μετάλλαξη ε, το Flams Belang, το κόμμα μου, δεν είναι αντίθετο προς την πρόοδο, αλλά ε, δεν θα πρέπει να είμαστε ε, όμοιροι στα χέρια των πολιεθνικών. Υπάρχει δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να απαγορεύουν την καλλιέργεια, να την περιορίζουν, αλλά όχι το εμπόριο ή την εισαγωγή. Και αυτό είναι διπλή επιβάρηση και διπλό μειονέκτημα. Δεν μπορούν οι αγρότες να τα καλλιεργούν, αλλά να τα εισάγουν επιτρέπεται τα κράτη-μέλη και οι φορολογούμενοι καταναλωτές αγοράζουν πιο φτηνά εισαγόμενα προϊόντα. Γι' αυτό το λόγο, για να αποφύγουμε κάθε παρανόηση, καταψήφισα ε, το κείμενο και κάνω την παρούσα επεξήγηση ψήφου. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό τώρα ο κύριος Πόλτσα. Ε, Σας ευχαριστώ. Εγώ υποστηρίζω την συγκεκριμένη πρόταση απλά γιατί πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα μπορέσουν να ωφεληθούν από μια τέτοια πρόταση. Είναι μια πρόταση η οποία θα δώσει λοιπόν την δυνατότητα να μπει μια κάποια τάξη. Ε, γιατί μέχρι τώρα οι χώρες δεν ήταν σε θέση μόνες τους να περιορίσουν ή και να απαγορεύσουν πλήρως ε, νομίζω λοιπόν ότι ε, υπήρχε μια σύγχυση από τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις που είχαν γίνει πριν από το 2001 και γι' αυτό ακριβώς ε, οι ευρωπαϊκές αρχές θα είναι σε θέση να ελέγχουν τους κινδύνους τους οποίους δημιουργεί η καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων και έτσι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την αρχή της επικουρικότητας. Κυρία Χάρκεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ένα από τα θέματα που συχνά, για τα οποία συχνά αναρωτήθηκα ήταν αυτό που συζητάμε σήμερα και ο τρόπος που ψήφισα, υπέρ δηλαδή, νομίζω ότι αποτελεί ένα θετικό βήμα για την απάντηση. Η τωρινή κατάσταση είναι τελείω απαράδεκτη. Μπορούν να μηνυθούν χώρες κατά πολυεθν... από πολυεθνικές. Ενώ έτσι επιτρέπεται η μη καλλιέργεια τροποποιημένων, ακόμη και αν οι περισσότερες χώρες είναι υπέρ. Τώρα δεν υπάρχει πια αυτή η δυνατότητα μήνυσης κατά των χωρών μελών. Μπορούν να αποφασίσουν μόνες τους. Η Ιρλανδία αποφάσισε να απαγορεύσει τα τροποποιημένα. Μετά τη σημερινή ψηφοφορία πρέπει να δούμε τι θα γίνει γενικά με την καλλιέργεια των μεταλλαγμένων. Η κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν από τους πολιτικούς να λάβουν αποφάσεις και τώρα που υπάρχει μια γνωμοδότηση για τα μεταλλαγμένα αν θέλουμε να πάρουμε υπόψη μας το παράδειγμα της Ουγγαρίας θα αναγκαστούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε το θέμα, να τεθεί το θέμα της κατανάλωσης των μεταλλαγμένων που δεν είναι άμυρα κινδύνων. Ελπίζω έτσι να μπορέσει να αλλάξει το ισχύον σύστημα και να ενισχυθεί η θέση των χωρών μελών που θα μπορούν να επιλέξουν. Οι μεταλλαγμένοι οργανισμοί μέχρι τώρα διευθετούνταν κεντρικά και τα κράτη-μέλη δεν είχαν πολλές δυνατότητες παρέμβασης. Νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε χάρη στο συμβιβασμό αυτό να έχουμε μια μεγαλύτερη νομική ασφάλεια, ιδιαίτερα για τις χώρες που θέλουν να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν την καλλιέργεια των μεταλλαγμένων. Γιατί υπάρχει το ΕΦΣΑ λέει τη για να κάνει επιστημονικές νοματεύσεις. Η ασφάλεια λοιπόν για την κατανάλωση τροφίμων από τα ζώα και τους ανθρώπους είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό όπως και ανησυχητικό. Δεν πρέπει να βασιστούμε μόνο στο συνέστημα αλλά στη γνώση. Οι πράσινοι μας έδωσαν την εντύπωση ότι τα μεταλλαγμένα είναι κάτι το τελείως τεχνητό. Τα κράτη-μέλη μπορούν να μην τα δεχτούν αν και υπάρχει ο κίνδυνος κατακαιρματισμού της αγοράς. Πώς μπορεί αυτό να συνδυαστεί με την ενιαία αγορά. Αν υπάρχουν μεταλλαγμένα πρέπει να μπορούν οι καλλιεργητές να γνωρίζουν τι ισχύει για να πάρουν μια απόφαση τα κράτη. Η κυρία Μακλάρκιν. Σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα θέλουμε αποφάσεις οι οποίες να βασίζονται σε επιστημονικές κυρίως απόψεις. Η ψηφοφορία αυτή θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να πάρουν τις αποφάσεις τους και το Ηνωμένο Βασίλειο βλέπει ότι μπορεί να παίρνει αποφάσεις στον τομέα αυτό αντίθετα από την κατάσταση πριν. Είναι για επιστρο... Μιλάμε για επιστροφή εξουσιών στην χώρα μου. Ο κύριος Γούλφ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η συγκεκριμένη πρόταση ήταν μια ευκαιρία και μια δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την αρχή της επικουρικότητας και να ανακτήσουν εξουσίες για τα γενετικά τροποποιημένα. Είπατε, ακούσατε ένα μέλος της, των συντηρητικών να λένε ότι ήταν μια καλή πρόταση. Δεν ισχύει αυτό, δυστυχώς. 50 παράγραφοι επιβάλλουν στα κράτη-μέλη ε, να προσαρμόζονται και να υπακούουν πριν πάρουν την απόφαση αυτή. Για μια ακόμη φορά στην ουσία δείχνει πόσο απάτη είναι αυτό εδώ το σώμα και πόσο υπερβολικές αρμοδιότητες έχει. Δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε στους πολίτες της Ευρώπης την επιλογή στα τρόφιμά τους. Δεν υπάρχει σύστημα για επιμόλυνση και δεν υπάρχει δυνατότητα για τους Ευρωπαίους πολίτες να πούν όχι αν θέλουν ή ναι εάν το επιθυμούν. Ευχαριστώ κύριο Σκέλη ένα λεπτό. Κύριε Κέλλη. Έχετε δίκιο κύριε Γκίλ, έχετε εσείς το λόγο, ο κύριος Κέλλη αμέσως μετά. Ο Βρετανικός τύπος και πάρα πολλοί βουλευτές λέγουν ότι αυτή η πρόταση θα επιστρέψει αρμοδιότητες και εξουσίες στην κυβέρνησή μας. Δεν είναι σωστός όμως, κάνω τίτλος, δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να απαγορεύουν την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και αυτό ισχύει πάντα εδώ στο Κοινοβούλιο. 50 από τις τροπολογίες ομαδοποιήθηκαν. Βλέπουμε εδώ ότι η τροπολογία 20 που πράγματι επιστρέφει αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη στην ουσία εξασθένησε από τις υπόλοιπες και γι' αυτό ακριβώς στήρισα στάση αποχής. Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ ψήφισα υπέρ της συγκεκριμένης πρότασης και με το πολιτικό μου κόμμα, το, την πολιτική μου ομάδα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ε, ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει και πράγματι ένα μεγάλο ποσοστό των βουλευτών, ε, το 70% υπερψήφισαν τη συγκεκριμένη πρόταση. Αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό, γιατί πράγματι δίνει την δυνατότητα ε, στα κρατημέλη να πάρουν τις αποφάσεις που θεωρούν καλύτερες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Στην χώρα μου, στην Ιρλανδία, ε, είναι πολύ καλή μια τέτοια δυνατότητα και την χρειαζόμασταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα κράτη-μέλη μπορεί να πάρουν διαφορετικές αποφάσεις αν το επιθυμούν. Παρ' όλα αυτά θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν τις επιλογές τους και αυτό είναι ένα σημείο προόδου ε, αν και δεν είναι κάτι εύκολο. Ο κ. Τσαμπάσκι, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπερψήφισα εγώ την πρόταση, διότι τη θεωρώ λογική. Και οι νέε ρυθμίσει είναι και λογικές, είναι και αυτό που χρειαζόμαστε. Στη Βουλγαρία ο κόσμος δείχνει μεγάλη καχυποψία στην καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων και απέναντι στα προϊόντα που προκύπτουν από τι καλλιέργειε αυτέ. Και με την παρούσα έκθεση δεν ε, προβλέπεται τίποτα για το εμπόριο και για την κυκλοφορία των προϊόντων στην αγορά. Το μόνο που αφορά η πρόταση είναι η καλλιέργεια, ο περιορισμός και η απαγόρευσή της. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις σχετικά. Στη Βουλγαρία οι περισσότεροι πολίτες είναι αντίθετοι με τις καλλιέργειες γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και εγώ τους υποστηρίζω και απευθύνω έκκληση σε Κομισιόν και Συμβούλιο να διευρύνουν τα δικαιώματα των κρατών μελών και να παίρνουν και την απόφαση ε, όχι μόνο για την καλλιέργεια αλλά και για την κυκλοφορία στην αγορά και τις εισαγωγές και, την μεταποίηση στο έδαφος τους. Κόμπο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή ψηφίζαμε. Δεν ψηφίζαμε αν μπορεί η Μεγάλη Βρετανία ε, ε, να καλλιεργεί ή να μην καλλιεργεί ε, μεταλλαγμένα. Μία τροπολογία ήταν μεταξύ 52 που το επέτρεπε, τα υπόλοιπα ήταν ακριβώς το αντίθετο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αποφασίζει. Η Βρετανική Βουλή και μόνο η Βρετανική Βουλή θα πρέπει να λαμβάνει τέτοιου είδους αποφάσεις για γενετικά μεταλλαγμένες καλλιέργειες. Το UKIP Ε, είναι αντίθετο ε, με ε, την πρόσβαση των αλλιέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα, κοντά στα νυχτά του Ισνήσου Μαγιώτ. Αυτό το θεωρούμε σε Ιχέλες επίσης. Το θεωρούμε ε, απεικιοκρατία και είναι πραγματικά πάρα πολύ ε, βλαβερό. Ο κύριος Χάναν, παρακαλώ. Όταν μιλάμε για τις κλιματολογικές αλλαγές σε αυτήν εδώ την αίθουσα, ακούμε συνέχεια ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να λατρεύουμε τις επιστημονικές συνενέσεις. Αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν λοιπόν αυτό το επιχείρημα, όταν ερχόμαστε στο σημερινό θέμα, ξαφνικά αλλάζουν άποψη δεν μιλάμε για επιστημονική συνένεση αλλά για τα αισθήματά τους. Εν στη δημοκρατία έχουμε ε, και ο καθένας μπορεί να λειτουργεί είτε εγκεφαλικά είτε συναισθηματικά. Μπορεί κάποιοι να πιστεύουν ότι αυτό δεν είναι πολύ λογικό αλλά εντάξει ο καθένας μπορεί να έχει και τις προκαταλήψεις τις οποίες θέλει είναι λάθος να επιβάλλει κανείς τα γενετικά τροποποιημένα σε κάποιον που δεν τα θέλει όπως και να απαγορεύσει σε κάποιον να τα προμηθεύεται εφόσον επιθυμεί να το κάνει. Γι' αυτό λοιπόν ας προχωρήσουμε σε λύσεις με τους εθνικούς μας τρόπους και διαδικασίες και όχι να προσπαθούμε να συνενέσουμε 600 εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Ο κύριος Άγνιου ένα λεπτό. Βλέποντας το θέμα φαίνεται εύκολο. Έχετε μια ευκαιρία να ξαναγυρίσουν αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη. Από την άλλη όταν το βλέπει κάποιος πιο προσεκτικά βλέπουμε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπλέκεται σε όλες τις φάσεις πολύ περισσότερο από όσο γίνεται σήμερα. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς στηρίσαμε στάση αποχές και θα έπρεπε όμως να ψηφιστεί η τροπολογία 20 γιατί αυτή πράγματι επέστρεφε αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη αλλά δυστυχώς την κατάπιανε οι υπόλοιπε τροπολογίες. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε οι χώρες οι οποίες δεν θα καλλιεργήσουν αν θα απαγορεύσουν στους καταναλωτές τους να τα καταναλώνουν. Αυτό θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ περίεργο ε, κάποιοι να μην έχουν την δυνατότητα να βρουν τρόφιμα λόγω της συγκεκριμένης ρύθμισης. Ο κύριος Φίντς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αποχή ψηφίσαμε, εμεί ζητώ συγγνώμη, <laughs> διάβαζα λάθος γραμμή στο κείμενό μου. Ε, εμείς είμαστε όλοι υπέρ του επαναπατρισμού των εξουσιών. Το πρόβλημα είναι οι τροπολογίες, όπως πάντα είναι αντιφατικές. Το τελικό πρόβλημα ποιος είναι. Στην αλήθεια, στην πραγματικότητα, όλα αυτά θα τα καταστήσει περιτά και θα τα καταργήσει η συμφωνία TTIP. Ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνονται οι επεξηγείς ψήφου. Έχω μια ανακοίνωση να σας κάνω. Ο πρόεδρος έλαβε από τις αρμόδιες